Σας παρακαλώ να καθίσετε κυρίες και κύριοι. Η διακοπή σαν την 12η Φεβρουαρίου ε, περίοδο συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επαναλαμβάνεται. Στο πρακτικό και τα κείμενα που εγκρίθηκαν σε εκείνη την περίοδο συνόδου είναι διαθέσιμα. Υπάρχουν ενστάσεις.